πέρυσι Η Κομισιόν ζήτησε το λόγο. Κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν βέβαια από την ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για λίγα λεπτά μονάχα που θα λάβει το λόγο η Κομισιόν, αλλά επειδή έχουμε πολλές ψηφοφορίες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συζήτηση. Σας παρακαλώ και πάλι να καθίσετε και να υπάρξει και κάποια ησυχία στην αίθουσα. Κύριε Ρεν, έχετε το λόγο. Thank you. Thank you, President. Uh, Honorable. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σε συμφωνία με την Προεδρία του Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής θα ήθελα να κάνω μια δήλωση εξ ονόματος της Κομισιόν για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για την Ελλάδα. Για να σας ενημερώσω και να στηρίξω την πολιτική σας στήριξη για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, για να διευκολυνθεί η επόμενη εκταμίευση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος για την Ελλάδα. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας καταλήξαμε σε μια συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού ε, της ε, Τρόικας και των ελληνικών αρχών. Η συνεδρίαση του Eurogroup ε, που ξεκίνησε τρίτη βράδυ μέχρι τετάρτη πρωί ε, σημείωσε ουσιαστική πρόοδο προς μια συμφωνία για το θέμα της Ελλάδας αν και δεν καταλήξαμε σε οριστικό συμπέρασμα αυτή τη φορά. Σημαντικό είναι πως το Eurogroup αναγνώρισε πως οι ελληνικές αρχές είχαν ε, εφαρμόσει επιτυχώς ε, όλες ε, τις προαπτούμενες δράσεις που είχαν συμφωνηθεί με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ. Κατά το οποίο βεβαίως δείχνει πολύ σημαντική προσπάθεια από πλευράς Ελλάδας. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις για να συγκροτηθεί μια πιο αποτελεσματική φορολογική διοίκηση. Αυτό έχει κρίσιμη σημασία γιατί βεβαίως ε, η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών ε, είναι και θέμα δημοσίων οικονομικών αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε τον μύθο πως ε, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην Ελλάδα. Και αυτή η εντύπωση βεβαίως είναι άδικη και λανθασμένη. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ελλάδα έχει επιδείξει αποτελέσματα. Τώρα έχει φτάσει η ώρα οι Ευρωπαίοι και οι διεθνείς εταίροι της Ελλάδος να κάνουν και αυτοί αυτό που τους αναλογεί. And uh, Και για να γίνει αυτό, το Eurogroup, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να συμφωνήσουν σε μέτρα αξιόπιστα για να ξαναγίνει βιώσιμο το χρέος ε, της Ελλάδας. Οι συζητήσεις ε, της Τρίτης μας έφεραν πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι σαφές πως ε, τα μέτρα αυτά δεν σημαίνει πως τα επόμενα χρόνια δεν θα επανεξεταστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και δεν αποκλείεται να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις όταν αυτές καταστούν αναγκαίες ε, ανάλογα με τις μελλοντικές εξελίξεις και την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα. Συμπερασματικά λοιπόν, ελπίζω πως ε, όλοι θα επανέλθουν στις Βρυξέλλες την επόμενη Δευτέρα με το απαραίτητο επικοδομητικό πνεύμα και θα ξεπεράσουν την καταστρεπτική νοοτροπία των κόκκινων γραμμών. Ειλικρινά δεν βλέπω κάποιον λόγο για να μην κλείσει το πακέτο και να σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα η οποία εμποδίζει την ε, επιστροφή της ε, ανάπτυξης και των επενδύσεων στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ελλάδας και σας διαβεβαιώ πως οι υπηρεσίες μου εργάζονται στο μέγιστο για να συμβεί αυτό και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε αυτή την ουσιαστική σημασία συμφωνία για την ευρωπαϊκή οικονομία και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Ρεν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος μου ζήτησε να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ερχόμενη Κυριακή είναι η διεθνή ημέρα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα όμως αυτή η βία στον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζει κοινωνικά